D'accord D'accord. Chers collègues, je vous invite à gagner votre... Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui étais responsable du... Μέχρι τώρα εγώ έφταιγα για την καθυστέρηση, αλλά από εδώ και πέρα εσείς θα φταίτε για οποιαδήποτε παρατέρω καθυστέρηση. Καθίστε λοιπόν για να μην καθυστερούμε άλλο και να μπορέσουμε να κηρύξουμε την έναρξη της συνεδρίασής μας. Πρόκειται για μια έκτακτη συνεδρίαση που έχουμε σήμερα το βράδυ. Πρώτα απ' όλα, η μερίσια διάταξη εγκρίνεται ή έχετε παρατηρήσεις. Εγκρίνεται λοιπόν. Δεν έχω ανακοινώσεις να κάνω. Και όσον αφορά τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 25 η 26ης Ιανουαρίου και τη 28ης Φεβρουαρίου, εγκρίνονται όσοι έχουν. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, ούτε ζητάτε κάποια διόρθωση. Καλώς. Οπότε, φτάνουμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε πρώτα ε, τροποποίηση για τον καθορισμό του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σας υπενθυμίζω ότι η ψηφοφορία αυτή είναι μια συνολική ψηφοφορία, ενιαία. Πρόκειται για ένα αδιέρετο σύνολο. Πρόκειται λοιπόν για ένα σύνολο που ψηφίζεται ενιαία μαζί. Συνεπώς, ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Θα κάνουμε πρώτα μία δοκιμή για να δοκιμάσουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δοκιμαστικά λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. 25 ψηφίζουν. Άλλος ένας πρέπει να ψηφίσει. Ένας από εσά δεν ψήφισε, ενώ έχει βάλει την κάρτα. Α, εντάξει, τώρα ψήφισε. Καλώς. Οπότε, Φτάνουμε στην ε, ψηφοφορία αυτή καθεαυτή τώρα που μας προτείνουν οι εισηγητές μας Γιάνν Όλμπριχτ και Ιζαμπέλ Τομά. Είπαμε ότι πρόκειται για νέα ψηφοφορία για τον ε, κανονισμό. Κύριε Όλμπριχτ, παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν είναι εδώ κυρία Τομά. Έχουμε τις τεχνικές πληροφορίες τώρα όσον αφορά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Μπορούμε δηλαδή να ψηφίσουμε στην Επιτροπή με την ενιαία ψηφοφορία, αλλά ίσως στην Ολομέλεια να χρειαστεί να ψηφίσουμε δύο φορές. Είναι οι κανόνες του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, η ψηφοφορία που κάνουμε τώρα, τεχνικά μιλώντας, μπορεί να μην είναι ταυτόσιμη με την ψηφοφορία που θα κάνουμε στην Ολομέλεια. Σήμερα είναι 9, ενώ μπορεί στην Ολομέλεια να έχει χωριστεί το κείμενο του κανονισμού αφενός και μετά να έχουμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. σε ευχαριστούμε για τη διευκρίνηση αυτή. Θέλουμε να υπάρχει συνοχή μεταξύ του κανονισμού και της ψηφοφορίας. Καλό θα ήταν λοιπόν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την Ολομέλεια να εμπνευστούν από τη δικιά μας ε, λογική επιχειρηματολογία και να υπάρξει μια ενιαία ψηφοφορία εφόσον πρόκειται για ένα σύνολο. Ο κανονισμός είναι μαζί με τις δηλώσεις ένα ενιαίο σύνολο. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε διαβάθμιση και να ψηφίσουμε χωριστά τον κανονισμό και χωριστά τις δηλώσεις. Είναι σαν να χάνεται το μήνυμά μας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω και θα το φροντίσετε κι εσείς στις ομάδες σας, έτσι όπως εκπροσωπούνται στη διάσκεψη των πρόεδρων, να επιμείνουν στον πρόεδρο να υπάρξει και στην Ολομέλεια ενιαία ψηφοφορία, όπως θα έχουμε και εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Λοιπόν, Παρακαλώ, κυρία Γαζαζαμπάλ. Θέλω να ψηφίσω. Δεν ήθελα να πω τίποτα. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίζουμε συνεπώς. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Συγχαρητήρια λοιπόν στους συνεισηγητές μας. Ήταν μεγάλη διαδρομή και περίπλοκη. Τα καταφέραμε όμως. Ερχόμαστε τώρα στην κινητοποίηση του περιθωρίου για τις απρόβλεπτες ανάγκες. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες που θα ψηφίσουμε. Τροπολογία αριθμός 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, Ρίτετε. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 3. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σύνολο τώρα της έκθεσης, υπέρ παρακαλώ. Α, ηλεκτρονικά πρέπει να ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες. Εγκρίθηκε 24 ψηφί υπέρ, 1 κατά και 3 αποχές. Συνεχίζουμε. Έκθεση Καρδιαζαβάλ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για τη χορήγηση εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για κάλυψη ζημιών από χρηματοδοτικές δραστηριότητε εκτός της Ένωσης. Έχουμε μακρύ κατάλογο ψηφοφοριών. Συμβαστική τροπολογία Α πρώτα απ' όλα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 62. Εδώ βλέπετε κάτι που θα ξαναβρούμε πολλές φορές. Λοιπόν, 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. τροπολογία 13 καταπίπτει, γιατί καλύπτεται από την 62. Τώρα, τροπολογία 12, υπέρ, κατά, αποχές, θα παληθεύσουμε. Γιατί δεν είναι ξεκάθαρο το πώς ψηφίζετε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, 16 κατά. Τροπολογία 67. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, Δεν είναι ξεκάθαρο. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται 14 κατά και 11 υπέρ. Αυτή ήταν η 13. 14 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ντε δέλτα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, 4 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις Απορρίπτεται. 14 κατά, 13 υπέρ. Αυτή ήταν η 4. Τροπολογία 71. Τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ δεν καταλαβαίνω πώς ψηφίζετε. οπότε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 71. Πέρας τις ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 15 κατά 13 υπέρ. Τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 72 έχει αποσυρθεί. 73 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την 74. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται 14 υπέρ 12 κατά. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Α, συγγνώμη λέει ο πρόεδρος. Εδώ κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 3 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρα της φοφορίας. Απορρίπτεται. 15-15 το αποτέλεσμα. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 7. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 15-14. Τροπολογία 76. Καταπίπτει. Γιατί εγκρίθηκε 7. Τροπολογία 16 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 20. Κατά τμήματα. Υπήρχαν τρία, αλλά το πρώτο καλύπτεται από κάποια άλλη. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά, θα επαληθεύσουμε για το τρίτο τμήμα ηλεκτρονικά. Τροπολογία 23 23ο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. εγκρίνεται 14 υπέρ, 13 κατά. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 9 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 19 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 19. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της φοφορίας. Απορρίφθηκε 17 κατά 11 υπέρ. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κοιτάξτε να σηκώνετε το χέρι σας καλά για να καταλάβουμε. 20 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά γιατί δεν καταλαβαίνω. Συμφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 14 υπέρ 13 κατά. Τροπολογία 18. Υπέρ κατά, αποχές και εδώ είμαστε πραγματικά ίσα ίσα από την μια και από την άλλη. Λοιπόν, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίστε παρακαλώ για τη 18. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται 17 υπέρ 12 κατά. Η 79 καταπίπτει την ίδια με τη 18. Τροπολογία 17 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω, λας επαληθεύσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφοριες εγκρινεται εγκρίνεται 15-13. Τροπολογία 10. 23, 24 και 25. Μαζί όλες αυτές. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τροπολογία 82 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 82 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίπτεται. 16 κατά, 14 υπέρ. Τροπολογία 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίας. Εγκρίνεται 17 υπέρ, 13 κατά. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 14 υπέρ, κατά, Εγκρίνεται νομίζω, αλλά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 17 υπέρ 13 κατά. Τροπολογία 23. Αν εγκριθεί θα σηκωνευτεί με τη 14. 23 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται. 86 υπέρ, να ελέγξουμε θέλετε. Ωραία, θα ελέγξουμε για τα 15 λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα της φοφορίας Απορρίπτεται 15-15 το αποτέλεσμα. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 16 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. Εγκρίθηκε. 18 υπέρ 12 κατά. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για τη 17. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτεται. 14 υπέρ 16 κατά. 91 και 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Η 94 καταπίπτει. Ναι. Όχι, αν εγκριθεί 92, οπότε 94 ψηφίζουμε υπέρ. Όχι, καταπίπτει μου λένε. Ωραία, καταπίπτει. 92. Και αυτή καταπίπτει. 24 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της Εγκρίθηκε 15 υπέρ, 12 κατά. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 96 καταπίπτει ή όχι. 96 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Οπότε ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε 17 υπέρ 13 κατά. 21 υπέρ. Α, όχι, λάθος λέει ο πρόεδρος. Καταπίπτει ή όχι. καταπίπτει. Γιατί 96 εγκρίθηκε. Καταπίπτει 21 λοιπόν. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική Β υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, όχι, 22 τροπολογία, 22 λέει ο πρόεδρος. Αλλά διορθώνει, συγγνώμη. Συμβιβαστική σε γάμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάλι 24. Της άφετ αυτή τη φορά υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 14 κατά 13 υπέρ. Συμβαστική α. Υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 131 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 της ΔΕΒΕ και 30 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται νομίζω αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 29 και την 30 λοιπόν μαζί ψηφίστε πέρας της ψηφοφορίας απορρίφθηκαν 16 κατά 13 υπέρ Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 133 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 134. 32 της ΔΕΒΕ. 33 της ΔΕΒΕ. 135 και 30 αφέτ. Υπέρ παρακαλώ. Μαζί. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις φοφορίες. Απορρίπτονται 17 κατά 13 υπέρ. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 35. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες απορρίφθηκε. 16 κατά, 13 υπέρ. 136 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 της ΑΦΕΤ υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις τώρα. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία αριθμό 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω, αλλά σε επαληθεύσουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για την τροπολογία αριθμός 1. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίνεται 16 υπέρ, 14 κατά. 38 υπέρ. Α, όχι, καταπτύπτει γιατί εγκριθήκε Τροπολογία 1 της ΑΦΕΤ. Υπέρ παρακαλώ. Α, και αυτή καταπίπτει, λέει ο πρόεδρος. 2. ΔΕΒΕ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 2 της ΔΕΒΕ. Ψηφίστε. Πέρες της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 16 υπέρ 14 κατά. Τροπολογία αριθμός 3. Κατά τμήματα. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 3. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε 17 κατά, 13 υπέρ. Τροπολογία αριθμός 1 της ΙΝΤΑ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία αριθμός 1 της ΕΝΒ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά.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 Πέραση της προφορίας Απορρίφθηκε 17 κατά 13 υπέρ. Τροπολογία 3 Τη ΣΥΝΤΑ υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 3 της ΑΦΕΤ υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 45 και 46 μαζί υπέρ κατά Αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία 5 της ΔΕΒΕ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της ΔΕΒΕ υπέρ. Κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε για την 6 της ΔΕΒΕ ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε 15 υπέρ 13 κατά. 4 αφετ υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε 4 της αφετ. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοβορίες. 16 κατά 14 υπέρ απορρίφθηκε. 5 αφέτ υπέρ. Δεύτερο τμήμα, γιατί το πρώτο εγκρίθηκε στα πλαίσια κάποιου συμβασμού. Δεύτερο τμήμα της 5 λοιπόν, της ΑΦΕΤ υπέρ, κατά. Θα επαληθεύσουμε. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 5 της ΑΦΕΤ, εξωτερικών υποθέσεων. Πέρας της Απορρίφθηκε 16 κατά 13 υπέρ. Τροπολογία 8. Δεύε υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 4. Τη σύντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50 και 9 μαζί. Υπέρ. Κατά. Δεν τα χέρια, βλέπω. Ωραία. Ηλεκτρονικά λοιπόν θα ψηφίσουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίφθηκε 17 κατά 13 υπέρ. 5 είναι υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 10 της ΔΕΒΕ υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 10 της ΔΕΒΕ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της προφορίας. Εγκρίθηκε. 17 υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 6 της ΑΦΕΤ και τροπολογία 6 της ΣΥΝΤΑ, που είναι οι ίδιες. Α, καταπίπτουν. 51 τότε. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2 NV υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 11 της ΔΕΒΕ υπέρ, κατά, αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 11 λοιπόν μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά πέρα της φοφορίες. Εγκρίθηκε 17 υπέρ, 14 κατά. Τροπολογία 7 είναι τα υπέρ. Α, καταπίπτει. Τροπολογία 7, αφέτη υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ. Α, καταπίπτει. γιατί εγκρίθηκε η 7 πριν. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 της ΑΦΕΤ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, συγγνώμη, τροπολογία 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 12 της ΔΕΒ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 8 είναι υπέρ, κατά, αποχές, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 8 της ΙΝΤΑ. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. 16 υπέρ, 13 κατά. Τροπολογία 9 της ΑΦΕΤ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 ίντα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε 16 κατά 14 υπέρ. Αυτή ήταν η 58. Τώρα τροπολογία 10 αφέτ υπέρ 10 λοιπόν υπέρ κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. 10 της ΑΦΕΤ. Ψηφίστε. Πέρας της απορρίφθηκε. 18 κατά 13 υπέρ. 10 ίντα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 ίντα υπέρ. Κατά. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά για την 11 της ίντα. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε 17 κατά 11 υπέρ. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Και τώρα ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία επί της ε, τροποποιημένης πρότασης της Επιτροπής με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 28 υπέρ 3 κατά. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε και για την ε, εντολή έναρξης διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Πάλι με ονομαστική ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίας. Οπότε εγκρίθηκε η εντολή. 28 ψήφι υπέρ, 2 κατά. Συγγνώμη που τόσο συχνά χρειάστηκε να προσφύγω στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά ήμασταν τσιματσίμα βλέπετε στο αποτέλεσμα κάθε φορά. Και τώρα ερχόμαστε στην έκθεση Γκάρδια Ζαμπάλ. Πρόκειται για την ε, εγγύηση και τις εξωτερικές δράσεις. Έχουμε την τροπολογία αριθμός 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ίντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 καταπίπτει 5 καταπίπτει επίσης εκτιμώντας 2 τοπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, εκτιμώντας 4 τοπολογία 1 υπέρ κατά εγκρίνεται εκτιμώντας 5 τροπολογία 2 υπέρ έχει καταπέσει. Εκτιμώντας 5, τροπολογία 1, ίντα, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Εκτιμώντας 5, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τώρα, για την ε, πρόταση της Κομισιόν όπως τροποποιήθηκε, με ονομαστική κλίση, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Και για την εντολή διαπραγματεύσεων με ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπέρ 27 ψήφοι, δύο αποχές, δύο μάλλον κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Γκουαρδιαζαπάλ. Nous avons des transferts, des virements. Έχουμε τώρα μεταφορές. Κύριε Γκάγερ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχει προχωρήσει αρκετά η ώρα, θα είμαι σύντομος. Τρεις μεταφορές στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Πρόκειται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ξηρασίας και την εκδίωξη ανθρώπων λόγω των δράσεων του Μπόκο Χαράμ σε σημεία της Αφρικής. Διαβάζουμε επίσης για την Ιεμένη. Τα χρήματα λαμβάνονται από το αποθεματικό επιγουσών αναγκών και ανέρχονται συνολικά 135 εκατομμύρια στις υποχρεώσεις και 105 στις πληρωμές θεωρώ ότι η δαπάνη αυτή είναι σκόπιμη και χρήσιμη. Ανησυχώ κάπως διότι με αυτά τα υψηλά ποσά εξαντλούμε περίπου το 1 τρίτο του εν λόγω αποθεματικού. Ίσως λοιπόν ε, να αντιμετωπίσουμε κάποια σπάνιδα μέσων, κονδυλίων δηλαδή, μέχρι τα τέλη του έτους. Πάντως, εν τέλει, η σύστασή μου είναι αποδοχή. Ευχαριστώ και γενικέ Εισηγητά. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Θέτω σε ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έγκριση της μεταφοράς. 3, 4 και 5. Έναρξη της ψηφοφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται. 20 ψηφοί υπέρ, 2 κατά ο κύριος Τάραντ για τους άλλους τομείς. Α, εσείς, εσείς κυρία Χαουταλά, ωραία. Έχετε το λόγο, αντικαθιστάτε τον κύριο Τάραντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι ο κύριος Τάραντ κολλείεται σήμερα για αυτό τον εκπροσωπό. Προτείνει δύο μεταφορές. Μία που αφορά την βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο από το 1201 βασική μισθή να αυξηθούν οι δαπάνες του 1406 contract workers, συμβασιούχοι εργαζόμενοι, σε σύνολο 100.000 ευρώ. Ο κ. Τάραντ επίσης προτείνει και μια δεύτερη μεταφορά στην κατηγορία αυτή για την ομάδα στρατηγικών επικοινωνιών της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Πρόκειται για 330.000 ευρώ από το 3004, κονδύλιο 3004, άλλα διοικητικά κόστη αντιπροσωπιών και να μεταφερθεί στο 2210 τεκμηρίωση και έξοδα βιβλιοθήκης. Προτείνει εδώ 190.000 ευρώ και επίσης σχετιζόμενο με αυτό ...2.213 ενημέρωση δημοσίου, εκεί να αυξηθεί κατά 140.000 ευρώ πάλι για να ενισχυθεί η ομάδα που κάνει στρατηγική επικοινωνία της Υπηρεσίας Εξωτερικών Δράσεων. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσει σα. Έχετε ερωτήσεις αγαπητοί συνάδελφοι. Όχι. Άρα θα τοποθετηθείτε τώρα πρώτα για το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν απαιτείται όμως ψηφοφορία. Αν δεν έχετε ενστάσει, μπορώ να θεωρήσω ότι εγκρίνεται η πρόταση. Μάλιστα. Για την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων έχετε ενστάσει για τη μεταφορά που προτάθηκε, όχι. Έχει καλώς εγκρίνονται λοιπόν οι δύο μεταφορές πιστώσεων. Έρχομαι στην κυρία Χολμάιερ και στον οργανισμό Frontex. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ε, ευχαριστώ που δίνετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ο Frontex ως γνωστόν αποκτά περισσότερο προσωπικό μέχρι το 2020. Προστίθεται χίλιοι συνεργάτες στον οργανισμό αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση στα γραφεία δεν αρκεί πλέον, ο χώρος δηλαδή των γραφείων. Γι' αυτό και προβλέπεται στο υφιστάμενο ήδη κτίριο της BNP Paribas να μισθωθούν και άλλοι όροφοι μέχρι ότου να μπορέσει ο Frontex να μετακομίσει σε ιδιόκτητο κτίριο γραφείων που προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2024. συνολική αύξηση 2,238 εκατομμύρια. Σχεδόν 600.000 ανά έτος. Αυτό, αλλά δεν χρειάζεται εδώ έγκριση, γι' αυτό έχω συντάξει γνωμοδότηση μαζί με τον κύριο Χόφμαν, όπου κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό το μεταβατικό κόστος. Δηλαδή θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος δύο ετών, όπου ενδέχεται να επικαλύπτονται κόστη δύο κτηρίων. Γι' αυτό και ζητούμε μεταβατική περίοδος να διαμορφωθεί όσο γίνεται συντομότερη για να εξοικονομηθούν δαπάνες που μπορεί να φτάσουν και τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Και ζητούμε από τον Frontex να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην συμβεί αυτό. Ποια είναι η πρότασή σας πιο συγκεκριμένα. Η δική μου πρόταση είναι να εγκριθεί η γνωμοδότησή μου που υποχρεώνει τον Frontex να ψάξει να βρει άλλον ενοικιαστή, ο οποίος θα αναλάβει το κτίριο, και αυτή την υποχρέωση θα πρέπει να την εκπληρώσει ο Frontex το συντομότερο δυνατό, μόλις θα γνωρίζει δηλαδή πότε θα εξέλθει από το κτίριο, ώστε τα, το μεταβατικό κόστος να ισούται με το μηδέν. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Έχετε ερωτήσεις ή σχόλια. Θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν την γνωμοδότηση της κυρίας Χολμάιερ. Ψήφι υπέρ, με το χέρι. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές. Η γνωμοδότηση σας εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ολοκληρώσαμε εδώ την ψηφοφορία. Τον λόγο θα δώσω στον κύριο Γιάνν Όλμπριχτ για τα θεμελιώδη στοιχεία της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μετά το 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την γνωμοδότηση που συντάσσουμε για την Επιτροπή Περιφερειών, μάλλον Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ρέτζι, του Κοινοβουλίου. Δηλαδή τα θεμέλια της πολιτικής συνοχής. Ο γνωμοδότηση που συζητάσουμε για λογαριασμό τη Ρέτζη. Και επειδή υπάρχει, υπάρχουν τεχνικοί λόγοι, ορισμένα στοιχεία περιλαμβάνονται στη γνωμοδότηση και ορισμένα από τα στοιχεία θα προσθεθούν ω τροποποίηση λόγω του περιεχομένου τη γνωμοδότηση. Επειδή στη γνωμοδότηση αναφερόμαστε μόνο στα δημοσιονομικά στοιχεία της, μελλοντική πολιτικής συνοχής, γι' αυτό ορισμένα στοιχεία τα οποία μάλιστα τονίζω εδώ, ιδίως ότι το μερίδιο της πολιτικής συνοχής στον νέο προϋπολογισμό θα πρέπει να παραμείνει ως ποσοστό για την συνολική πολιτική, είναι αναγκαίο να βρεθεί μια διαστατική λύση που να αποφύγει νέο backlog, νέα καθυστερούμενα. Και θα πρέπει να ενισχυθεί η ευκαμψία και να αντιμετωπιστούν οι νέε προκλήσει στη διάρκεια τη δημοσιονομική προοπτικής. Γι' αυτό το αποθεματικό πολιτική συνοχή μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή που θα πρέπει να εξεταστεί. Να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να αντιδρούμε για να τα χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα αυτά για νέε προκλήσει. Μία από τι τροποποιήσεις λέει ότι αν πρόκειται για μακροπρόθεσμη πολιτική το ζήτημα τη διάρκεια πρέπει να ληφθεί υπόψη. αυτό θα πρέπει να προστεθεί, ε, μάλλον αυτό είναι στη γνωμοδότηση και αυτό που θα προστεθεί στο επόμενο στάδιο θα είναι να υπάρχει ε, μια ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών εργαλείων και των επιχορηγήσεων. Να υπάρχει δηλαδή μια καθαρή εργαλειοθήκη η οποία θα επιτρέπει να αντιλαμβάνονται οι δικαιούχοι ποιοι μηχανισμοί χρησιμοποιούνται για ποιο σκοπό. Εγώ προτείνω να εξετάσουμε τους νέους ενδεχόμενους δείκτες πέραν του ΑΕΠ για την πολιτική συνοχή. Πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα και νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί με καθαρό τρόπο πριν να δώσουμε τελική μορφή στην δομή της επόμενης πολιτικής συνοχής, γιατί έχουμε και νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, τα δημογραφικά και άλλα που πρέπει να την υπόψη και όχι μόνο το καθάριστο εθνικό προϊόν. Ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Σιγητά για την ε, τοποθέτησή σας που θα υποβληθεί τώρα σε ανταλλαγή απόψεων. Και πρώτη κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Επισημαίνω ότι η μεγαλύτερη απλοποίηση θα ήταν να έχουμε μια σταθερότητα. Όχι κάθε φορά από ένα δημοσιονομικό πλαίσιο σε άλλο να έχουμε αλλαγές διότι κάθε 7 χρόνια τα ξαναβάζουμε όλα επιτάπητος, υπάρχει μια επικάλυψη και τελικώς βεβαίω όλοι καταθέτουν τα όπλα. Εγώ θα κάνω μια τροπολογία, θα ζητάξω μια τροπολογία που θα γράψω ακριβώ αυτό. Πρόεδρος, νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, διότι όταν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέλαβε τα καθήκοντά του, διαπίστωσε ότι υπήρχε ένα έλλειμμα επενδύσεων και πρότεινε ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων για να ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Είδαμε όμως και την έναρξη του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ να πάσχει από μια μεγάλη αδράνεια δύο-τριών ετών, διότι οι επιχειρηματίες δεν επωφελήθηκαν από το νέο πρόγραμμα. Αν υπάρχει λοιπόν μια σταθερότητα στο νέο πρόγραμμα, αυτό θα επιτρέψει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες επενδύσεων. Άλλα σχόλια δεν βλέπω, ευχαριστώ πολύ. Οπότε, για την έκθεση αυτή, το χρονοδιάγραμμα, τροπολογίες, θα πρέπει να κατατεθούν έως τις 31 Τρίτου στις 11 το πρωί, ψηφοφορία στις 25 Τετάρτου, στην Επιτροπή δηλαδή, η επί της ουσίας αρμόδια Επιτροπής, στις 18 Μαΐου ψηφίζει δηλαδή. Το λόγο λαμβάνει πάλι ο κύριος Ολμπριχτ. για τα διαθωτικά ταμεία και το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, και την αύξηση των υποχρεώσεων. Εσείς κύριε Σιγητά. Μου επιτρέπετε, Πρόεδρε. Το θέμα αυτό αφορά την ορατότητα, την ε, διάδοση των επιδόσεων του ε, ε του Είναι γνωμοδότηση, συγγνώμη, ΕΣΥΦ, προς την ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και εν γέννη οι επιδόσεις ε, δεν είναι γνωστές για πολλές ε, ευρωπαϊκές χώρες και όταν βλέπουμε τα λαϊκιστικά κινήματα ακριβώς εκεί ποντάρουν στον κόσμο που δεν γνωρίζει ποιες επενδύσεις προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμού τα στοιχεία ε, από δημοσιονομικής άποψης, όχι μόνο δηλαδή χρήματα για τεχνική αρρωγή, αλλά κυρίως ε, και πάνω απ' όλα χρήματα για την επικοινωνία, ώστε πραγματικά να είναι ορατά τα όσα γίνονται, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε ορατότητα για τα αποτελέσματα αυτά. Μπορούμε να συζητήσουμε όσο θέλουμε το δημοσιονομικά, αλλά να κάνουμε καλή δουλειά, τελικά να μην γίνονται γνωστά τα αποτελέσματα. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να δούμε κάποια ειδική αρρωγή για την επικοινωνία οι Ευρωπαίοι πολύ συχνά διαμαρτύρονται ότι δεν γνωρίζουν τι γίνεται από ευρωπαϊκέ επενδύσει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εμεί δεν κάνουμε και πολλά ώστε να τα γνωστοποιήσουμε τα όσα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ για τι παρατηρήσει σα και αυτό ισχύει ε, και σε άλλου τομεί και όχι μόνο σε αυτά τα διευθυντικά και επενδυτικά ταμεία. Ο κ. Κέλμελ. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, αφού ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Όλμπριχτ. Συμφωνούμε και νομίζω ότι θα πρέπει βέβαια να ενστερνιστούμε και εμείς αυτό που λένε. Δηλαδή κάνε το καλό και μίλα για το καλό που έκανες. Αλλά πρώτα βέβαια πρέπει να αποκαταστήσουμε και την σαφήνεια, την καθαρότητα για το ποιο πράγμα έχουμε κάνει, τι έχουμε κάνει. Ιδίω τα τελευταία ένα-δυο χρόνια υπάρχει ένα έλλειμμα εκεί. Βλέποντας έγινε πάλι μια συζήτηση. Όλα αυτά τα έλα διαφόρων διαρθωτικών προγραμμάτων που ωστόσο έρχονται και επανέρχονται στις, στους ίδιους στόχους στήριξη μικρομεσών επιχειρήσεων και άλλα σχετικά. Αυτό τελικώς είναι αδιαφανές. Γι' αυτό νομίζω ότι ένα μεγάλο βήμα προς περισσότερη διαφάνεια θα είναι, θα κερδιθεί αυτό δηλαδή, εάν τα καταφέρουμε να μην υπάρχουν παράλληλες κινήσεις στήριξης ενισχύσεων για τα ίδια έργα. Να υπάρχει ένα πρόγραμμα που θα περιλαμβάνεται ενός έργου. Ευχαριστώ κύριε Μαλετίτσου. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το θέμα της επικοινωνίας και της ορειτότητας ΚΑΠ συνήθως έρχεται στο τέλος του προγράμματος της Επιτροπής μας, του Κοινοβουλίου και δεν έχουμε ποτέ αρκετό χρόνο να το συζητήσουμε, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γιατί όταν για παράδειγμα βλέπει κανείς το εύση και την ορατότητα αυτού και πόσο ο αντιπρόεδρος Κατάινεν έχει κάνει τη γύρα της Ευρώπης για να παρουσιάσει το εύση και από την άλλη πλευρά το, τα ΕΣΥΦ, τα Ευρωπαϊκά Διευθυντικά και Επενδυτικά Ταμεία που έχουν τόσα χρήματα διαθέσιμα για πολλά και διάφορα προγράμματα και συγκρίνουμε πόσο και αν ε, κάναμε προσπάθεια για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής, δεν κάναμε και πολλά. Πρέπει να γίνουν περισσότερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω πως τώρα έχουν συστήσει μια νέα μονάδα με μόνο αυτόν, αυτό έργο αλλά ε, αυτή η μονάδα δεν έχει αρκετό διοικητικό δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να βοηθήσουμε ώστε να φτιαχτεί αυτή η δυνατότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ στο επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στην, και χρήμα στην αρατότητα των ε, ταμείων αυτών. Ευχαριστώ συνάδελφε, ο κύριος Όλμπριχτ για να κλείσουμε. Πολύ σύντομα να πω πρόεδρε ο κύριος Κόλμα έχει απόλυτο δίκιο. Βεβαίως δεν θέλουμε να κάνουμε προπαγάνδα. Θέλουμε να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες. Και αυτές οι πληροφορίες θα έπρεπε να μοιράζονται σε αυτό που θα θέλαμε να κάνουμε στο σχεδιασμό και δεύτερον τις πληροφορίες και το τι κάνουμε στην πράξη που είναι διαφορετικές πληροφορίες και το τρίτο κομμάτι τα αποτελέσματα τι έγινε στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα αυτά ε, συνήθως έρχονται μετά από κάποια χρόνια θα πρέπει να είναι αυτό σαφές γιατί συχνά κάνουμε τη δημοσιοποίηση, δίνουμε δημοσιότητα στο τι κάνουμε, αλλά δεν τονίζουμε επαρκώς τα αποτελέσματα. Όταν λοιπόν ε, καταρτίζουμε μια πολιτική επικοινωνιακή, θα πρέπει να είναι σαφέ. Είναι ένα όνειρο αυτό. Α φανταστούμε, α ονειρευτούμε ότι μια μέρα των ημερών θα έχουμε ένα ταμείο για όλα. Τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία δεν είναι για τα πάντα, αλλά σε ελπίσουμε πω κάποια μέρα θα γίνει μια απλοποίηση και θα έχουμε ένα μόνο ταμείο. Έχω κι άλλο ένα όνειρο. Α ε, φτιάξουμε ένα καθαρό, ε, μια, μια ξεκάθαρη εργαλειοθήκη να έχουμε το τι κάνουμε, το τι έχουμε, ποιο πρόγραμμα έχουμε για ποιο αποτέλεσμα. Το ΕΦΣ έχει πολύ καλά αποτελέσματα, το ΕΣΥΦ επίση, αλλά δεν έχουμε καλή ε, δημοσιοποίηση αυτών. Πολύ περίπλοκο είναι αυτό, γιατί εγώ βλέπω ε, συγγνώμη που μακρηγορώ και έτσι αργεί η συνεδρίαση, αλλά ε, γίνονται πολύ περίπλοκες επιχειρήσεις και μετά λέμε να, αυτός εδώ είναι ο χρηματοδότης, ο δωρητής, ο χορηγός και η Ευρωπαϊκή Ένωση για ποσά που είναι πολύ μικρά. Και τελικά οι διάφοροι φορεί είναι πολύ πονηροί γιατί καταφέρουν να συγκεντρώσουν χρήματα από παντού, αλλά δεν αξιοποιεί αυτό δεν δίνει μάλλον αξία στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι ένα σωρό εχορηγή και τελικά η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν γίνεται αρκετά ε, ορατή. Και αυτό είναι ζήτημα. Επιπλέον, η πρόσβαση σε αυτά τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι τόσο περίπλοκη, γιατί υπάρχουν τα προγράμματα που τα ορίζει η Κομισιόν. Στη συνέχεια έρχεται το κράτος και θέτει τους δικούς του όρους και δημιουργεί και, άλλη, ε, ε, και άλλες επιπλοκές και μετά επειδή οι περιφέρειες κάνουν το, ε, την, την μοιρασιά βάζουν και αυτοί κάτι ακόμα από γραφειοκρατία και πραγματικά γίνεται καυκική κατάσταση. Η απλοποίηση θα βελτιώσει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί φαίνεται ως ένα τέρας περιπλοκότητας και γραφειοκρατίας. Εφόσον άλλος δεν θέλει το λόγο, να διευκρινίσω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι 12 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών στις 11 Μαΐου και τέλος θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια στις 12 Ιουνίου. Συνάδελφοι, η επόμενη μα συνεδρίαση θα γίνει στι 3 Απριλίου στι 8 το βράδυ μέχρι, 20, μέχρι τις 9.30 Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα ε, στο Στρασβούργο, στα διάφορα δεν έχουμε τίποτα. Πέρα στη συνεδρίαση, σας ευχαριστώ και καλό σας βράδυ.